Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ καθίστε. Χαιρετίζω τους πολυπληθείς συναδέλφους που είναι παρόντες. Καλώς ήρθατε. Στη συνεδρίασή μας τόσο νωρίς το πρωί χαιρετίζω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρώτο θέμα της της διάταξης είναι οι δηλώσεις.